πρώτα από την συνάδελφο Εύα Ζολή. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχει ένα σημαντικό νέο το οποίο δεν καλύφθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισητισμού χρειάστηκε να μειώσει κατά 20% τα τρόφιμα τα οποία πηγαίνουν προς την ε, Συρία ακριβώς επειδή δεν υπήρχε απαραίτητη χρηματοδότηση. Στην πράξη, αυτό όμως έχει να κάνει, μάλλον στην πράξη οδηγεί σε δραματικές συνέπειες ακριβώς επειδή δεν υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κοινωνικός προπολογισμός πιέζονται πάρα πολύ από δημοσιονομικής πλευράς και όντως ο Ευρωπαίος πολίτης επιβαρύνεται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και από τις πολιτικές λιτότητος που έχουν, υποβληθεί, έχουν επιβληθεί με συγχωρείτε, από πολλές κυβερνήσεις. Εννιά όμως Ευρωπαίους τους 10 συνεχίσουν να πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την, την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Ευρωπαίοι πολίτε, παρά την κρίση αυτή παραμένουν αλληλέγγυοι. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να ακούσουν τους πολίτες αυτούς. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε διάφορες αποστολές σε διάφορες περιοχές του κόσμου που πλήττονται από τη φτώχεια την ανέχεια. Κεντρική Αφρική, Συρία, Σουδάν, χώρες στις οποίες έχουμε πολύ σημαντικές σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες συνεχίζονται μάλιστα. Πώς είναι ποτέ δυνατόν να αποδεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σημαντικός δωρητής και ενισχυτής, μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει ένας αποστασιοποιημένος ε, παράγοντας για τις ε, ανθρωπιστικές αυτές κρίσεις χώρες ήταν σε θέση να συμμετέχει. Πώς μπορούμε να αποδεχθούμε το ότι μολονότι υπάρχουν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν θίξει το ζήτημα αυτό, καταλήξαμε τελικά με το να εγκρίνουμε έναν μειωμένο υπερπολογισμό. Το να μειώσουμε τώρα τις δράσεις αλληλεγγύης απέντη στους γείτονές μας, αυτό θα έστελε ένα απέσιο μήνυμα. Το μήνυμα μιας ανεδιπλωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρώπης η οποία είναι αδιάφορη για τον υπόλοιπο κόσμο. Η ελληνική λοιπόν στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι πολύ σημαντική και η ελληνική εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ουσία η ελληνική αυτή. Αποτελεί μέρο του κοινού μα DNA. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτού που έχουν ε, ανάγκη τη βοήθειά μα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατόν να καταφέρουν να εγκρίνουν έναν διορθωτικό προπολογισμό. Τα κράτη-μέλη επίση θα πρέπει να δείξουν το απαραίτητο θάρρο διότι ο εταίρος μας στο Ισραήλ για πολλωστή φορά ουσιαστικά καταστρέφει στην δυτική όχθη πάρα πολλά προγράμματα ή προϊόντα τα οποία έχουν ε, πραγματοποιηθεί, υλοποιηθεί χάρη στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε πλέον τις καταστροφές αυτές χωρίς συνέπεια, χωρίς κυρώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από τη στάση του Ισραήλ και πέρα από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες που έχουμε τη χώρα αυτή, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταγγείλουμε μια παραβίαση ακόμα του ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς ανθρωπικού δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να πιέσουμε το Ισραήλ να καταβάλει τις απαραίτητες αποζημιώσεις όχι μόνο για τις καταστροφές της 28ης Απριλίου, αλλά όλα αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν προκύψει ως ζημία εξαιτίας των καταστροφών που έχει προωθήσει το Ισραήλ, ιδίω όσον αφορά κάποια προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ε, για την περίοδο 2001-2011. 30 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό. Τα 30 εκατομμύρια ευρώ είναι η χρηματοδότηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι το Δεκέμβριο προκειμένου να στηρίξει τα θύματα της κρίσης που πλήττει τη Συρία. 30 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό αυτό το οποίο κάθε εβδομάδα χρειαζόμαστε στην Συρία προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες της χώρας αυτής καθώς επίσης και τους Σύρους πρόσφυγες στις όμορες χώρες. Τα 30 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό αυτό που δίνουμε, που δώσαμε τουλάχιστον το 2013 στο Αφγανιστάν ως ανθρωπιστική βοήθεια. Αλληλεγγύη λοιπόν υπευθυνότητα αλλά και αυστηροί κανόνε. Αυτό ακριβώς πρέπει να επιδείξουν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζολή. Το λόγο έχει ο συνεισηγητή μα, ο κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Ζολή μας ανέφερε τις δραματικές ε, συνέπειες της ε, έλλειψης ε, πόρων. Διέτασε ότι αφορά την επισητιστική και την αναπτυξιακή βοήθεια προς ε, χώρες που είναι τέρι μας. Δυστυχώς, παρόλο ότι το θέμα αυτό είναι, παρόλο η κατάσταση είναι δραματική και το θέμα είναι επίγον, εμφανίζεται σε όλα τα κεφάλαια των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το τέλος, στο τέλος του 2012, για πρώτη φορά, ε, διαπιστώσαμε μια πρώτη κρίση πιστώσεων πληρωμών που ε, μας οδήγησε να εκτελέσουμε τον προπολογισμό του 2012 με ένα μικρό έλλειμμα. Ξεκινήσαμε το 2013 με υπόλοιπα πιστώσεων του 2012 που έπρεπε να πληρωθούν το 2013 και παρά τον ένα γενναιόδωρο διορθωτικό πρόσθετο προπολογισμό μάλλον ε, είχαμε το τέλος του 2013 να φτάνει με μια έλλειψη πιστώσεων ε, που ξεπερνούσε τα, με ένα έλλειμμα πιστώσεων πάνω από 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Για πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει το 2013. Τώρα, στο μέσο του 2014, πάλι έχουμε κίνδυνο να μας, λείψει, να μας λείψουν ποσά. Έχουμε 700 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιμα σε σχέση με το, με το όριο, ε, με την οροφή του 2014. Συζητήσαμε με τον κύριο Λεβαντόφσκι και με την Επίτροπο Γεώργεβα και μας έδωσαν και δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη μας για όλες τις πληρωμές που είναι δυνατόν να γίνουν σήμερα για επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως, αυτές οι πληρωμές Αυτά τα εμβάσματα προέρχονται από γραμμές του υπερπολογισμού που γνωρίζουμε ότι θα είναι ελληματικές στο τέλος του χρόνου. Ε, συνήθως η μεταφορά ποσών γίνεται από γραμμές που υποχρησιμοποιούνται προς γραμμές του υπερπολογισμού οι οποίες εξαντλούνται. Όμως αυτή τη στιγμή ε, κόβουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Ε, όλο αυτό το σύστημα θα μπορέσει να εφαρμοστεί μόνο αν το Συμβούλιο αποφασίσει ένα πρόσθετο προϋπολογισμό στο μέσο του χρόνου ή εν πάση περιπτώσει πριν το φθινόπωρο. Ο κ. Λεβαντόφσκι θα μας ενημερώσει. Όμως ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το Κοινοβούλιο θα βρίσκεται σε παρένθεση για τέσσερις μήνες. Γιατί δεν θα μπορεί να ε, ψηφίσει από μόνο του ε, ένα πρόσθετο το συμπληρωματικό προπολογισμό. Ε, θα πρέπει να περιμένουμε. Από την άλλη μεριά <laughs> θα πρέπει να αφήσουμε ε, την, τον προπολογισμό σε τάξη τώρα που τελειώνουμε τη θητεία μας πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε αρκετά ποσά έτσι ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες πληρώμες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ. Του Συμβουλίου θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα. Ε, Madame le Président, ε, le Conseil est pleinement conscient ε, des problèmes το Συμβουλίο γνωρίζει το πρόβλημα των πιστώσεων πληρωμών για την εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανησυχίες τις οποίες ε, εκφράστηκαν από τον κύριο Ζόλη και τον κύριο Λαμασούρ. Ε, από πλευράς Επιτροπής Προπολογισμού και Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ήδη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα αυτό στον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό που έλαβε χώρα στις 2 Απριλίου. Η συνάντηση αυτή μας επέτρεψε να καθορίσουμε δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε τα χρηματοδοτικά προβλήματα που επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μας έδωσε μια αρχική αντίδραση για την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών, για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υποβάλλοντας δύο προτάσεις μεταφορών πιστώσεων. Το Συμβούλιο έκανε μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο προτάσεις μεταφορών αντιμετωπίστηκαν ως το ταχύτερα. Και με χαρά σας ενημερώνω ότι από την αρχή της τρέχουσας ε, εβδομάδας, μετά από την έγκριση στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας τον, τη Δευτέρα, η Κομισιόν είχε δυνατότητα να εγγράψει τα ποσά που απαιτούνται στην, ε, στις ανάλογες γραμμές του προπολογισμού. Εάν αυτές οι συμπληρωματικές ε, πιστώσεις δεν επαρκέσουν για να, καλύψουν, για να καλύψουν τις ανάγκες ε, των γραμμών αυτών αργότερα φέτος, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για ανακατανομή των πιστώσεων ή αν δεν επαρκούν για ένα σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Θέλω να σας διαβεβαιώσω το Συμβούλιο θα σεβαστεί πλήρως τη διατύπωση και το περιεχόμενο της κοινή δήλωσης για τις πιστώσεις πληρωμών που συμφωνήθηκε από τα τρία θεσμικά μας όργανα πέρυσι τον Νοέμβριο στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2014. Σύμφωνα με τη δήλωση λοιπόν αυτή, το Συμβούλιο θα αντιμετωπίζει ταχαίως οποιαδήποτε αίτηση για μεταφορά πιστώσεων πληρωμών συμπεριλαμβανομένων και μεταξύ διαφόρων τομέων του προπολογισμού. Επίση θα καταλήγει σε θέση για έναν ενδεχόμενο διορθωτικό προπολισμό όσο το δυνατόν ταχύτερα για να αποφευθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση και έλλειψη στις πιστός πληρωμών. Παράλληλα, καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να προκαταλάβω τη θέση που μπορεί να λάβει το Συμβούλιο για οποιαδήποτε συγκεκριμένη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Τώρα θέλω να πω λίγα λόγια για το προτινόμενο σχέδιο ενίσχυσης προς την Ουκρανία της Ένωσης. Είναι ένα θέμα που βεβαίως απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να υποστηρίξει το λαό και την κυβέρνηση της Ουκρανίας στις προσπάθειές τους να σταθεροποιήσουν τη χώρα και να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό το Συμβούλιο καλωσορίζει τη συνολική προσπάθεια υποβολής πακέτου ενίσχυσης που υπέβαλε η Κομισιόν και είναι δεσμευμένο να διασφαλίσει την εφαρμογή του. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ε, συμπληρωματική πίεση στις ε, πιστώσεις ή πληρωμών του ενωσιακού προπολογισμού κατά το τρέχον έτος. Ο τριμερής διάλογος για τον προπολογισμό στις 2 Απριλίου ήταν ευκαιρία για τα τρία θεσμικά μα όργανα να ανταλλάξουν απόψεις και από αυτού του θέματος. Η Επιτροπή, εν τω μεταξύ, έχει αναλάβει μια πρώτη σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το Συμβούλιο υποσχέθηκε να αντιδράσει ταχαίως. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταλήγοντας υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή έχει την ε, ε, αρμοδιότητα πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή λοιπόν πρέπει να μα υποβάλει προτάσει για ανακατανομή στον προπολογισμό ή για σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Το Συμβούλιο από την πλευρά του δεσμεύεται να εξετάσει η αδίποτε τέτοια πρόταση ταχαίω και να καταλήξει σε θέση ως να το πιο σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κούρκουλα. Τώρα ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Όντως η διαχείριση του προπολογισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια διαχείριση ελλημάτων τελικά. Είναι μια διαχείριση μειωμένων πόρων. Έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό έχει να κάνει με το ότι προβλέπονται συνεχώς λιγότερες ε, πληρωμές, λιγότερες πιστός πληρωμών σε σχέση με τις εκτιμήσεις που γίνονται. Αυτό το είδαμε το 2012, 2013 και 2014. Συνεπώς γνωρίζουμε πώς, είναι, πώς έχει η κατάσταση, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε σε μια πρώτη φάση τον εφαρμοστικό προπολογισμό και συνέχεια ακολουθεί συνήθω ένας διορθωτικός προπολογισμό σε σχέση με τις πραγματικέ ανάγκες, τα πραγματικά δεδομένα τα οποία μας υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Γιατί ακόμα και σε περίοδο κρίσης πρέπει κανείς να καταβάλει και να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς. Αυτό ισχύει ακόμα και για τα νοικοκυριά. Το 2014 ήταν και θα είναι μια δύσκολη χρονιά, καθότι βρισκόμαστε 9 δισεκατομμύρια κάτω σε σχέση με τα επίπεδα που είχαμε στον προηγούμενο προπολογισμό. Θα έχουμε λοιπόν ανεπάρκεια πόρων, ανεπάρκεια πόρων σε όλε τι γραμμέ του προπολογισμού, όχι μόνο στην εξωτερική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περίπου 20 δισεκατομμύρια τιμολόγια τα οποία δεν μπορούμε να καταβάλουμε όσον αφορά την πολιτική συνοχή και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί συνεχή προβλήματα στην εφαρμογή του προπολογισμού του 2014. Βέβαια αντιδρούμε και στις επιστολές αλλά και στα προφορικά ερωτήματα της κυρίας Ζολή και του κύριου Λαμασούρ και συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση στον τομέα των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, χρησιμοποιώντας επίσης τα μέσα τα οποία έχουμε χάρη στη συνθήκη και χάρη στο δημοσιονομικό κανονισμό. Και αυτό το είδαμε επίσης στα πλαίσια της κοινή δήλωσης που έχουμε για τις πιστώσεις πληρωμών και παραθέτω ότι το ανώτατο επίπεδο πληρωμών θα γίνει και βάση του περιθωρίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται χρησιμοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα μέσα ευελιξίας που προβλέπονται στη συμφωνία της, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέτρο του δυνατού θα χρησιμοποιήσει όλα τα νέα μέσα τα οποία προβλέπονται από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν είχε γίνει και στο παρελθόν. Ξέρετε ότι το 2013 είχαμε κινητοποιήσει επιπλέον 54% πιστώσεις πληρωμών όσον αφορά την πολιτική ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά. Ποια είναι η εργαλειοθήκη που έχουμε ε, στη διάθεσή μας. Πρώτον, η εποπτεία, η παρακολούθηση. Αλλά ουσιαστικά αυτό μας βοηθάει μόνο να εντοπίσουμε τις ανάγκες. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε κάποια μέτρα πρόληψης, χρησιμοποιούμε τα προληπτικά αυτά μέτρα, στα πλαίσια, για παράδειγμα, της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπου έχουμε μειώσει τα επίπεδα προχρηματοδότησης για κάποιους διεθνείς οργανισμούς. Τρίτον, τρίτο εργαλείο, οι μεταφορές, οι μεταφορές πιστώσεων πληρωμών. Ήδη μία θα γίνει με τη μορφή γεφυροποίησης προς την, προς την πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας και ιδίως όσον αφορά το μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ξέρετε ότι ορισμένε γραμμέ του προπολογισμού καταβάλλονται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο του έτου, αλλά παρόλα αυτά εμεί πρέπει να βρούμε ήδη εκ των προτέρων τα κονδύλια εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε αυτέ τι γραμμέ του προπολογισμού. Ήδη από τώρα πρέπει να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε δηλαδή κάποια ποσά. Επίση χρησιμοποιούμε το μέσο έκτακτη ανάγκη και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο αργότερα στο έτος χρησιμοποιούμε στο δυνατόν περισσότερο τη δυνατότητα ανακατανομή των πιστώσεων. Στο δεύτερο ήμιση του έτου γνωρίζουμε καλύτερα τι μπορεί να ανακατανεμηθεί. Και τέλο, χρησιμοποιούμε το μέσο του διορθωτικού προπολογισμού. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε μεταγενέστερο επίση στάδιο του έτου. Βλέπουμε πολλέ φορέ ότι μπορεί ο προπολογισμό και ο διορθωτικό προπολογισμό να μην αρκεί και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και όλα τα μέσα ευελιξία τα οποία τώρα προβλέπονται. Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, συμφωνώ με τι ερωτήσει τι οποίε θέσατε. Πρόκειται για μια βοήθεια η οποία πραγματικά σώζει ζωέ. Άρα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την πολιτική αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα. Όσον αφορά τώρα την Ουκρανία, ναι, πάλι πρέπει να βρεθούν επιπλέον πιστώσει στα πλαίσια του προπολογισμού 2014-2020 για τα 11 αυτά δισεκατομμύρια 1,4 έχει να κάνει με επιδοτήσεις, ενώ το υπόλοιπο έχει να κάνει με δάνεια τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια των εγγύσεων του κοινοτικού προπολογισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε τουλάχιστον τα ποσά αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινητοποιηθούν το συντομότερο δυνατό εξαιτία των ραγδαίων αυτών εξελίξεων στην Ουκρανία. Συνάδελφο Πρέντα έχει πρώτο το λόγο για δύο λεπτά. Mulțumesc, um, doamna președinte. Vreau să salut dezbaterea de astăzi pe tema deficitului Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι για αυτή την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σήμερα περί έλλειψης πιστώσεων πληρωμών για τη χρηματοδότηση εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Γιατί, ξέρετε, η επόμενη συνοδός μας θα είναι το καλοκαίρι. Οπότε το θέμα αυτό είναι πολύ επίγον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη. Θα ήθελα να ξαναμιλήσω για την κλίμακα του προβλήματος. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό είναι το 50% του συνολικού ετήσιου προπολογισμού της ανθρωπικής βοήθειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 150 εκατομμύρια θα πρέπει να αναζητηθούν μέχρι το καλοκαίρι για να μην δημιουργηθεί κρίση πληρωμών, σύμφωνα με την ΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν σημαντικά ανθρωπιστικά προγράμματα σε χώρες που πλήττονται. Προφανώς σε περίοδους κρίσης ε, όλος ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περικόπτεται. Οπότε αυτό επηρεάζει και τις υπόλοιπες γραμμές του προπολογισμού, όχι μόνο αυτήν της εξωτερικής βοήθειας. Όμως υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι παράγοντες. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι διαφορετική φύσεως από τι άλλες, άλλες του προπολογισμού. Ε, πολλές ε, φορές ε, χρειάζεται να είμαστε πολύ ταχεί στην παρέμβασή μας ιδιαίτερα όταν έχουμε ξηρασίες, ένοπλες συγκρούσεις, πλημμύρες κλπ. Η Γενική Διαντσιέκο το 2013 μόνο βοήθησε 130 εκατομμύρια άτομα. Πίσω από τα νούμερα έχουμε πραγματικούς ανθρώπους στη Συρία, τον Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και τώρα στην Ουκρανία. Πρόκειται για ανθρώπους που βασίζονται στη βοήθειά μας. Τέλος, ε, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μία από τις ε, πιο δημοφιλείς δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι θέμα αξιοπιστίας μας. Ευχαριστώ. E e- Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε διάφορες ανθρωπιστικές αποστολές στις Φιλιππίνες, στον Νότιο Σουδάν, στην ε, Συρία. Και ορισμένες φορές ε, μας δίνει την εντύπωση ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Δεν υπάρχει συντονισμός. Ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναλάβει συγκεκριμένε υποχρεώσει χρηματοδότησης οι οποίε αυτή τη στιγμή ενδεχομένω να μην μπορούν να λεωποιηθούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα των πιστώσεων πληρωμών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχή μείωση τη βοήθεια που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πολύ συχνά αναφερόμαστε σε καταστάσει όπου διακυβεύεται ακόμα και η ίδια η ζωή των ανθρώπων. Αν μιλάμε αυτή τη στιγμή για να κατανομή στα πλαίσια του προπολογισμού, αυτό είναι μία μέθοδο, αλλά από μόνη τη δεν αρκεί. Γιατί ξέρετε ότι αναφερόμαστε σε γραμμέ του προπολογισμού που και αυτέ αργότερα μέσα στο έτο θα αποδειχθούν ελληματικέ. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο ποσό κονδυλίων προκειμένου να αποκριθούμε στι υποσχέσει μα. Και από την άλλη, προσπαθούμε να δώσουμε και χρήματα σε ακόμα περισσότερε χώρε, όπω για παράδειγμα στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τα κονδύλια αυτά να είναι διαθέσιμα. Η Επίτροπος Γεωργίευα έχει πει ότι αν μη τι άλλο θα πρέπει να μπορούμε χρηματοοικονομικά να καλύπτουμε τι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει. Κάθε φορά όμω που αναλαμβάνουμε νέε υποχρεώσει και δίνουμε νέε υποσχέσει, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Διαφορετικά οι υποσχέσει μα είναι εντελώ φρούδε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε επίση να εξασφαλίσουμε και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώ επίση και του Μέσου για την Ασφάλεια. Εδώ τα ποσά είναι πάρα πολύ ελληματικά. Πώ μπορούμε να αναλάβουμε δράση στα πλαίσια των μέσων αυτών, αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, αν δεν συνάπτουν τελικά λόγια και πράξει. Προσπαθούμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να ανακατανύμουμε κάπως τα ποσά και να παρουσιάσουμε εκ νέου κάποια προγράμματα τα οποία είναι ελληματικά. Και παράλληλα θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και την Ουκρανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αποκριθούμε στο αίτημα αυτό της Επιτρόπου Γεωργίευα για 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υπολείπονται στον κοινοτικό προπολογισμό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να έχουμε τα κονδύλια αυτά. Το κόστος των παρεμβάσεων δείχνει την σημασία του προβλήματος. Οι κρίσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, είναι ε, ε, πολύ πλατιές. Η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στον Νότιο Σουδάν, τη Σύρια, ε, καθιστούν απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφιερώσει μεγαλύτερα κονδύλια. Όμως ας είμαστε ρεαλιστές. Τα ποσά τα οποία απαιτούνται εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλά. 150 εκατομμύρια μέχρι τον Ιούνιο, συν 150 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι πρόσθετα ποσά τα οποία θα χρειαστούν για την ανθρωπιστική δράση το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλάβει τι ευθύνε του. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Όπω το έκανε και η Επιτροπή Προπολογισμών τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση με την πρώτη δόση των 150 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ε, ε, ε του δισταγμού των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα 400 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί μια εξαιρετική περίπτωση κατάσταση. Ε, ενώπιον σημαντικών κρίσεων είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στα θύματα ότι ε, έχουμε γίνει παρατηρητές ε, ανήμποροι, παρατηρητές τέτοιων καταστάσεων εξαιτία ε, ε, πόρων. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα αύξησης των ποσών. Ε, ε, τόση προσπάθεια όμως για μια απλή μεταφορά ποσών ε, πρόκειται για ασφαλώς για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά όλα αυτά έχουν σχέση με την διεθνή αλληλεγγύη. Ε, Ο συνάδελφος Πουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκι, Συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ που ως συγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Μηχανισμό για την Σταθερότητα και την Ειρήνη μπορώ να λάβω σύντομα το λόγο. Το πρόβλημα που έχει αναφερθεί ήδη εδώ για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας υπάρχει στον ίδιο βαθμό και στον τομέα για τον οποίο είμαι υπεύθυνο. Είναι βέβαια μικρότερα τα ποσά, αλλά είναι θεμελιώδη. Μας λείπουν 58 εκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου. Πρόκειται για προγράμματα που υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν να γίνουν λοιπόν σε 9 χώρες. Ουκρανία, Ιράκ, Γκάζα, Συρία, Ιράν, Σιέρα Σουδάν, Νότιο Σουδάν και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πρόκειται για ε, βασική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή η αντιμετώπιση σειράξεων και η πρόληψη σειράξεων και μάλιστα πολλές φορές ε, εμφυλίων σειράξεων και νομίζω ότι γελιοποιούμεθα αν δεν είμαστε σε θέση να δαπανίσουμε τα ποσά αυτά, να βρούμε τα ποσά αυτά και τονίζω ότι δεν πρόκειται για ανταγωνισμό, δεν αντιπαρατηθέμεθα προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Όχι, σαφώς όχι. Βεβαίω η ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται περισσότερο όταν ακριβώς δεν έχει υπάρξει πρόβληψη. πρόληψη. Συγγνώμη και η Βαρόνη Άστον ε, το έχει αναφέρει επανειλημμένα. Ε, ευχαριστώ για αυτά που υπόθηκαν και παρακαλώ συγκεκριμένα τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι να υπάρξουν τα φορές πιστώσεων και για το μηχανισμό για σταθερότητα και ειρήνη όπως ήδη το προτείνατε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ τον Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι είπε πριν από λίγο ότι ε, η έλλειψη πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ε, είναι μια πραγματικότητα αναπόφευκτη. Όμως στην πολιτική δεν υπάρχουν τέτοιες αναπόφευκτες πραγματικότητες, υπάρχουν επιλογές. Και οι επιλογές που έχει κάνει το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο για θέματα προπολογισμού είναι καταστροφικές ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να μπουν στη θέση κάποιου που μας ακούει και περιμένει απελπισμένα τη βοήθειά μας. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένα πολύ μικρό ποσό του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεύτερον, πριν από λίγο καιρό στην Επιτροπή Προπολογισμών ήρθε κάποιο από την Παλαιστίνη και μα ε, μίλησε για την δραματική κατάσταση που επικρατεί εκεί. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν μπορούν να περιμένουν την σύσταση του Κοινοβουλίου, ούτε την ε, αύξηση, ούτε την δράση της Κομισιόν του Συμβουλίου. Εκεί κάθε μέρα χάνονται ζωές θα αποκτήσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική εξωτερική πολιτική αποτελεσματική. Αν είχαμε τέτοιου είδους ε, πολιτική, ίσως αποφεύγαμε και την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Μιλούμε για την έλλειψη 150 εκατομμυρίων ευρώ αλλά θα πρέπει να καταγγείλω τους τελευταίους ε, μήνες ε, λέμε σε χιλιάδες ανθρώπους, ε, τους ζητούμε μάλλον από χιλιάδες ανθρώπους συγγνώμη για την έλλειψη αυτών των ποσών, για την έλλειψη νερού, φαρμάκων, καταφυγίων, ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή τη φορά μπορούμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί που υποχρέωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει συγγνώμη επειδή δεν έκανε το καθήκον της ό,τι αφορά τα, το, δεν έκανε το ανθρωπιστικό της καθήκοντα. Είναι οι εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών. Ε, τους προειδοποιώ ότι αυτό το κοινοβουλίο δεν θα ε, επιτρέψει στο Συμβούλιο να υπογράφει λευκές επιταγές για την Συρία, την Κεντροαφική Δημοκρατία κλπ. Γιατί κάθε φορά που αυτή η βοήθεια δεν δίδεται χάνουν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 150 εκατομμύρια, αλλά η τρύπα είναι 450 εκατομμύρια. Τι θα κάνει το Συμβούλιο για να πάψουμε να παίζουμε ρώσικη ρουλέτα τις ε, ζωές των ανθρώπων αυτών. Δεν θα το επιτρέψουμε ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Κορτέρ Λάστρα. Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε ακόμα πολύ δύσκολου καιρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν νομίζω ότι οι πιο φτωχοί θα πρέπει να φέρουν το βάρο. Η ανεπάρκεια αυτή κονδυλίων όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια ουσιαστικά βάλει και κατά μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στο μέλλον δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να χρηματοδοτούμε τις πολιτικές αυτές. Είμαστε πραγματικά σοβαροί όμως όσον αφορά τις θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν περικόπτουμε καταρχάς για τους ανθρώπους εκεί, πόρους από τους ανθρώπους εκείνους που χρειάζονται τους πόρους αυτούς. Ποιο μήνυμα ουσιαστικά στέλνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση προς το τέλος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κρίση στη Συρία. Αναφέρομαι και στι υποσχέσει που έχουμε δώσει προ τι χώρε εκείνε που δέχονται πρόσφυγε από τη Συρία. 9 εκατομμύρια. Θεωρώ πραγματικά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου είναι πάρα πολύ σημαντική. Προστατεύει άνδρε και γυναίκε ε, υποστηρίζει επίσης όλους τους υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα είναι η στιγμή πραγματικά να χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές αυτές. Μετά από 15 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά παίρνω για τελευταία φορά το λόγο. Ουσιαστικά θα ήθελα να πω προς ψηφοφόρους μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να σταθώ δίπλα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που υποστηρίζουν τους άλλου πολίτες. Η Ευρώπη μας θα πρέπει να Μάλλον πρέπει να υποστηρίξουμε την, Ευρώ... την Ευρώπη μας αυτή, η οποία θα πρέπει να βασίζεται προφανώς στη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Ουδής άλλος έχει ζητήσει τον λόγο για το Catch the Eye. Να ζητήσω λοιπόν από τον Επίτροπο Λεβαντός και να πάρει το λόγο. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος κυρία Πρόεδρε. Όντω, αντιμετωπίζουμε ανεπάρκειες και λήψεις στο σύνολο του κοινοτικού προπολογισμού. Το 2014 θα είναι ένα δύσκολο έτος όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, γιατί έχουμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από ό,τι είχαμε κατά την εκτέλεση του προπολογισμού 2013. Και προφανώς χρειαζόμαστε κονδύλια στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε εκατομμύρια ευρώ και εγώ δίνω αυτή τη στιγμή την υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο από τον δημοσιονομικό κανονισμό και από την συνθήκη προκειμένου να κάνουμε ό,τι δυνατό μέσω μεταφοράς πιστώσεων ή κατανομής πιστώσεων για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια αυτά. Χωρί όμω φρέσκο χρήμα δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλες αυτές οι υποχρεώσεις μας, δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλους τους λογαριασμούς του οποίους πρέπει να πληρώσουμε. Καταλαβαίνετε, τα κονδύλια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ιδίω όσον αφορά την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δηλαδή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη ανθρωπιστική τη δράση σώζει ζωέ. Θα κάνω κάθε τι το δυνατό, αλλά επαναλαμβάνω ότι χωρί επιπλέον κονδύλια, χωρί φρέσκο χρήμα, δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να βρεθούν επιπλέον πόροι μέσω, της, μέσω του νέου κοινοβουλίου. Ο κύριος Κούρκουλας έχει το λόγο εξ ονόματος Συμβουλίου. It is important to meet the European Union's budgetary needs, particularly in the area of humanitarian aid. We are committed to supporting this important policy under the heading 4 of the Multiannual Financial Framework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 γιατί ε, θα περάσει κάποιο διάστημα ε, μέχρι να υπάρξει ο επόμενος πρόεδρος στα ελληνικά. Είναι και για μένα, όπως και για τον συνάδελφο Μαρτίνεθ, Μαρτίνεθ η τελευταία φορά που προεδρεύω να... και είναι ιδιαίτερη διπλή χαρά μου που αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες θερμότατα για την ε, εξαιρετική συνεργασία. Ε, είμαι περήφανη και νομίζω ότι όλες μας και όλοι μας πρέπει να είμαστε περήφανοι που υπηρετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική θητεία και θα ήθελα επίσης ε, ως Ελληνίδα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ουσιαστική υποστήριξη και αλληλεγγύη που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Αντιπρόεδρος Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ που προείδρευε πριν από μένα, κατεβαίνουμε από το τρένο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά σε καμία περίπτωση δεν κατεβαίνουμε από το τρένο της Ευρώπης, το αντίθετο μάλιστα θα είμαστε στο πρώτο βαγόνι στην πρώτη γραμμή. σας ευχαριστώ πολύ και σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση θα διακοπεί μέχρι τις έξι που θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες.